ich erkläre die am. 12. September. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση που διακόπηκε στις 12 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Και... βεβαίως οι συνάδελφοι όπως είναι λογικό θα σιωπήσουν και θα επικρατήσει ησυχία. Αλλά στην ησυχία αυτή υπάρχουν κάποιες κραυγές. Κραυγές παιδιών που βλέπουν τους γονείς τους να πνίγονται. και φωνές γονιών που δεν μπορούν να σώσουν τα παιδιά τους. Φωνές ανθρώπων που χάθηκαν στη μανιασμένη θάλασσα παρά το ότι έβλεπαν τις ακτές της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Της Υπήρου στην οποία πίστευαν ότι θα βρουν προστασία και ελπίδα. είναι οι κραυγές των ανθρώπων που λίγο πριν φτάσουν στην ακτή της Ευρώπης έχασαν τη ζωή τους. Συζητάμε για αριθμούς. Ε, το πόσοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Ποιος θα λάβει ποιους και πόσους πρόσφυγες και πόσο κοστίζει. Συζητάμε για ξερές παραγράφους. Να μην είμαι κατάσταση η οποία είναι απίστευτη. Ότι οι ψαράδες που έσωσαν τους ανθρώπους θα τιμωρηθούν για βοήθεια, προς, ε, για βοήθεια σε παράνομη μετανάστευση. Τη στιγμή που η πλουσιότερη Ήπειρος του κόσμου Ναι, ε, βεβαίω είμαστε οι πλουσιότεροι ήπειρο του κόσμου, αλλά δεν είναι σωστά μοιρασμένο ο πλούτο, το ξέρουμε αυτό. Αλλά εμεί πολίτες σε σχέση με αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται είμαστε πλούσιοι, ισχυροί, ικανοί. Και αυτοί φεύγουν από την συμφορά τους για να βρουν εδώ πέρα προστασία και ελπίδα. Σε σχέση με αυτούς τους ανθρώπους είμαστε πλούσιοι και ισχυροί. Θα ήθελα να μιλήσουμε για παραγράφους στο πλαίσιο αυτό αλλά για τη δύναμή μας και τον ευρωπαϊκό πλούτο. Που παρόλες δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, πρέπει να αποτελεί για μας μια υποχρέωση. Υποχρέωση να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που ζητάν προστασία από μας. Ελπίζω το λεπτό υγιής για τα θύματα της ε, τραγωδίας της ε, Λαμπεντούζας θα αποτελέσει ίσως ένα σημείο καμπής στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ.